Κυρίες και κύριοι, άρχεται η συνεδρίαση. Η γραμματεία με πληροφορεί ότι πρέπει εγώ με τη σειρά μου να σας ενημερώσω πως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά. Λάβετε το υπόψη σας, αν και η συμπεριφορά σας ήταν πάντοτε εξαίρετη και άψογη. Στόχος της συνεδρίασης είναι αποκλειστικά η εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 191 του κανονισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια υποψηφιότητα. Ναι, υπάρχει υποψηφιότητα. Mr. Clint, please. Κύριος Κλίνθ. Micro. Κοιτάξτε, ω ε, συντονιστή ε, μέχρι σήμερα τη Επιτροπή των Φιλελευθέρων στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Επιθέσεων θα ήθελα να προτείνω Sharon Both, ε, την κυρία Sharon Both ω πρόεδρο αυτή τη Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και πρόθυμη να αναλάβει αυτή τη θέση που εκφράζει την διαθεσιμότητά τη. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Όχι, έχουμε μία μοναδική ε, υποψηφιότητα της κυρίας Σάρων Μπόλ, η οποία ζητάει το λόγο και της τον δίνω με πολύ χαρά. Ήθελα να κάνω μία δήλωση ε, πριν ανακοινώσετε τον ορισμό μου. Ε, με τιμά η υποψηφιότητα αυτή εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων. Παίρνω πολύ στα σοβαρά τον ρόλο της Προέδρου και γνωρίζω τις ευθύνε μου ενώπιον όλων των πολιτών. Για λόγους διαφάνειας και επειδή η Επιτροπή αυτή έχει αναλάβει το διάλογο με την Κεντρική Τράπεζα θα ήθελα να αναφέρω τη δική μου προσωπική θέση σχετικά με το ευρώ. Εγώ ήμουν και είμαι πάντοτε υπέρ του ευρώ και υπέρ της ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στη ζώνη του ευρώ. Αυτό το γνωρίζουν πολλοί από τους συναδέλφους μας που είναι παρόντες τώρα και ήταν και στην προηγούμενη θετία. Έχει καταγραφεί στα πρακτικά, αλλά θα ήθελα να το επαναδιατυπώσω σήμερα. Αυτή είναι και η θέση των φιλελεύθερων δημοκρατών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως ε, ε, ευρωβουλευτής ε, ανήκω στην ομάδα των φιλελευθέρων και ενστερνίζομαι τις θέσεις της ομάδας μου και σε ό,τι αφορά το θέμα του ρυθμιστικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα. Θα συνεργαστώ υπεκοδομητικά με την Επιτροπή του συντονιστέ και το Προεδρείο. Αυτή είναι, αυτός είναι ο ρόλος μου και αυτός είναι ο ρόλος οποιοδήποτε Προέδρου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νομισματικές υποθέσεις και το νομισματικό διάλογο είμαι και θα εξακολουθήσω να, και θα παραμείνω ε, δεσμευμένη και προσιλωμένη την ε, υπεράσπιση των συμφερών και αυτών των χωρών που είναι στο ευρώ και όλων των χωρών που επιθυμούν να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ. Έχουμε μια εξαιρετική υποψηφιότητα. Αυτή η δήλωση ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και εξαιρετική. Και αν δεν υπάρχουν άλλοι εξαιρετικοί υποψήφοι, θα προτείνα ε, να την εκλέξουμε δια voice. Εκλέγουμε την κυρία Σάρων Please, will you take the chair, please. Παρακαλώ, ελάτε να πάρετε τη θέση σας στο Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα έχω ε, να ακολουθήσω αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στον ε, διορισμό των αντιπροέδρων. Οπότε, θα ήθελα να ακούσω τις υποψηφιότητες για την θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Jean Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, επιτρέψατε μου να σα συγχαρώ πρώτο και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δήλωση που μόλι κάνατε. Ω πρώην και νέο ε, συντονιστή εξ ονόματο του ΕΛΚΑ, προτείνω για την Αντιπροεδρία την υποψηφιότητα του συναδέλφου Γκαρσία Μαργάλιο που, υπήρχε, που ήταν στην θέση σας μάλλον ε, πριν από σας. Thank Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Δεν βλέπω καμιά άλλη υποψηφιότητα, οπότε προτείνω να προχωρήσουμε στον διορισμό διαβοής. Ah, Ελάτε, περάστε. Ε, σειρά σας να κάνετε και εσείς δύο βήματα. Uh, Ωραία. για την θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Βλέπω τον κύριο Σκινά. Κυρία Μπόλς, κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην θέση αυτή. Ε, πολύ σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη τις ε, δηλώσεις σας. Ελπίζουμε πως θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση που περιγράψατε. Εγώ προσωπικά έχω την τιμή να ανακοινώσω την υποψηφιότητα του δεύτερου αντιπροέδρου ε, της κυρίας Αρλίν Μακάρθη που είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής. Την γνωρίζετε πολύ εδώ. Θα είναι μια, ένας πολύ καλός σύνδεσος μεταξύ της δουλειά που κάνουμε τώρα και είναι δική μας υποψηφιότητα από την πλευρά μας για τη δεύτερη Ευχαριστώ. Δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Διαβοής λοιπόν η Αλήν Μακάρθη ορίζεται ως δεύτερη διπρόεδρος. Um, um, η Αρλίν κάνει τώρα τα βήματα, τα δύο βήματα mm-hmm. και να ρωτήσω ποιες είναι οι για την τρίτη αντιπροεδρία. Ο κύριος Γκόζες και πάλι. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προτείνω για την τρίτη αντιπροεδρία τον κύριο Στόλοζαν. Uh, thank σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Περάστε. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ε, μετάφρασης, αλλά πρόκειται για εκλογή και όχι για διορισμό. Κάνουμε εκλογές τώρα και όχι διορισμούς. Πιστεύω ότι το σύστημα είναι να υπάρχει πρώτα μια υποψηφιότητα και μετά να εξετάζουμε άλλες υποψηφιότητες. Εγώ πάντοτε με πρότεινε κάποιος ως υποψήφιο πριν να είμαι υποψήφιος. Υπάρχει πρόταση υποψηφίων. Ε, λοιπόν, προτάσεις για αυτούς που μπορεί να εκλέξουμε ως τέταρτο αντιπρόεδρο. Ο κύριος Σκίνερ, σας ευχαριστώ. Και πάλι έχω την τιμή να ανακοινώσω την υποψηφιότητα του Έντουαρτ Σικ Κλούνα που είναι Μαλτέζος υποψήφιος από την αντιπροσωπεία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχει ιδιαίτερα προσόντα, είναι πρώην πρόεδρος της ε, Μαλτέζικης Αντίστοιχης Επιτροπής και της, της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Μάλτας και πιστεύω πως θα κάνει εξαίρετο έργο στην Επιτροπή μας. Σας τον συστήνω όλος ιδιαίτερος. Thank Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Ωραία λοιπόν, τότε μπορούμε να εκλέξουμε τον κύριο Σακλούνα διαβοής. Right. Um... Uh, Έχω κάποιες ανακοινώσεις ε, του Πρόεδρου. Η ημερομηνία της επόμενης συνεδρία της Επιτροπής θα είναι η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 12.30 και επίσης από τις 3 μέχρι τις 6.30 της ίδιας μέρας. Αυτά και τώρα ε, κυρίως το πέρα συνεδρία. Σας ευχαριστώ όλους.